Κάνετε μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δεν είναι πολύ εύκολο να παρακολουθεί κανείς τόση πολλή ώρα τις εργασίες μας και σας ευχαριστώ για αυτό. Λοιπόν, κλείνει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Το επόμενο θέμα είναι πλέον η έκθεση φύσας για την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Έχετε κύριε Σιγητά το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να σας συγχαρώ και εγώ για το νέο σα αξίωμα. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Βασιλείου και τους συναδέλφους στην Επιτροπή Πολιτισμού και του σκιώδης ηγητέ από τι πολιτικέ ομάδε για την πολύ καρποφόρα συνεργασία που είχαμε του τελευταίου μήνε. Σήμερα ο κόσμο του αθλητισμού πενθεί. Πενθεί για του νεκρούς σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αίγυπτο. Θα ήθελα να εκφράσω τη διδρυμίτα την καταγγελία μου και την καταδίκη μου και τα συλληπιτήριά μου προ τα θύματα και τι οικογένειε, των θυμάτων. Η έκθεσή μου μιλάει για τι συνεχείς επαφέ με τον κόσμο του αθλητισμού. Θέλουμε να ακούσουμε τις ανησυχίες τους και να δούμε για ποια θέματα ζητούν ε, την επέμβαση ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη της Λισαβόνα ε, ε, δημιούργησε επανάσταση για τον αθλητισμό γιατί για πρώτη φορά δημιουργεί στο άρθρο 165 μια νομική βάση για τον αθλητισμό. Και μάλιστα η πρώτη απάντηση στη συνθήκη ήταν ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Διάσταση του Αθλητισμού, που ακολουθεί τι οδηγίε τη Λευκή Βίβλου του 2007. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μία έκθεση πρωτοβουλία, δώσαμε απάντηση σε αυτή την ανακοίνωση. Και μάλιστα η έκθεση αυτή, με 28 ψήφου υπέρ και 2 κατά, εγκρίθηκε στην Επιτροπή Πολιτισμού. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημαντικά ορόσημα ε, για τον αθλητισμό που ήλθαν υπόψη στην έκθεσή μου. Καταρχήν, η αρχή της επικουρικότητας που αναγνωρίζει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και η αρχή της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 165 της Συνθήκης. Βέβαια, αυτή δεν είναι μια οικουμενική αρχή. Θα πρέπει να εξεταστεί και περιπτωσιολογικά να εγκρίνεται. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σεβαστούμε την αυτονομία των διαφόρων δομών διακυβέρνηση του αθλητισμού, που είναι το βασικό θεμέλιο τη οργάνωση του αθλητισμού. Θα ήθελα τώρα συντομία να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία τη έκθεση. Καταρχήν, ο εθελοντισμό η ανιδιοτελή συμμετοχή χιλιάδων πολιτών που εξασφαλίζει τη διοργάνωση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων ε, και θα πρέπει να υποστηρίξουμε ανεπιφύλακτα τον αθλητισμό. Δεύτερο, φαρμακοδιέγερση. Το ντόπινγκ είναι μάστιγα και για τον αθλητισμό και για την κοινωνία. Θα πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε τον κόσμο, να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη, να ε, κυνηγήσουμε τους ε, ε, λαθρεμπόρους και να επιβάλλουμε κυρώσεις, φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και το συμφέρον των αθλητών. Θα πρέπει να, να ε, ε, διώξουμε το λαθρεμπόριο ουσιών ντόπινγκ όπως διώκουμε και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Είναι σημαντική διαπαιδαγώγηση από την αρχή και συμπερίληψη του αθλητισμού από το δημοτικό η ζωή του αθλητή αργά ή γρήγορα τελειώνει. Είναι σημαντικό λοιπόν πέραν της αθλητικής σταδιοδρομίας να μπορεί ο αθλητής να παρακολουθήσει και διάφορα μαθήματα για να μπορέσει στη συνέχεια να ανακυκλωθεί. Άσχετα ε, από τον αθλητισμό έχουμε πολλές φορές ε, ρατσιστικές, ξενόφοβες ή ε, ομοφοβικές τάσεις και στον αθλητισμό. Θα πρέπει ε, αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουμε στις αθλητικέ εκδηλώσεις. Ο αθλητισμός έχει σημαντικά ωφέλη και για την υγεία, γιατί μειώνει και ταυτόχρονα μειώνει και τις ε, κρατικέ δαπάνες για την υγεία. Άλλωστε έχει και κοινωνικό ρόλο και εντάσσει καλύτερα στην κοινωνία τις πιο ευάλωτε ε, ομάδες όπως είναι οι κοινωνικά αποκλεισμένες, ομάδε οι ανάπηροι ή οι μετανάστε. Θα πρέπει να, να προστατεύσουμε τα στοιχήματα, αλλά να καταπολεμήσουμε τα παράνομα στοιχήματα και το στήσιμο των αγώνων. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα κυριότητας των οργανωτών ε, διαφόρων εκδηλώσεων και επίσης να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις για το στήσιμο αγώνων και τέτοιου είδους απάτες. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε τις αθλητικές εκδηλώσεις με περιφερειακό και κεντρικό τρόπο, ώστε να γίνει σαφής, καταχω... σαφής καταμερισμός και δίκαιος καταμερισμός του κέρδους του αθλητισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί όχι να μην έχουμε και ένα αθλητικό έρασμος και να προστατεύσουμε τον αθλητισμό ως τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα θέματα που αναλύονται στην έκθεση, για την οποία ζητώ την υποστήριξη σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην αρμόδια επίτροπο, την κυρία Βασιλείου. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα και εγώ να εκφράσω να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Και επίσης ε, ως επιτροπός αρμόδια για τον αθλητισμό δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για αυτά που συνέβησαν στην Αίγυπτο σήμερα. Για αυτό το λόγο ακριβώς λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε υπέρ του υγιούς τρόπου διεξαγωγής του αθλητισμού σε κάθε εκδήλωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή, τον κύριο Φίσας και τους κοιόντες εισηγητές για όλο το έργο τους και για την εξαιρετική έκθεση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση για τον αθλητισμό. Θα ήθελα να σημειώσω ότι με χαρά βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ανακοίνωσης του προηγούμενου Γενάρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις προτάσεις της έκθεσης. Δύο χρόνια μετά τη θέση σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας ε, εφαρμόζουμε μια συνεκτική ομάδα δράσεων στον τομέα του αθλητισμού βάσει προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Μετά από την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον Αθλητισμό και το σχετικό πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεσή του ολοκληρώνει ένα συνοπτικό πλαίσιο για την πολιτική, για τον αθλητισμό για τα επόμενα χρόνια. Να αναφέρω κάποιες πρωτοβουλίες εν συντομία, τις οποίες θα εκτελέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει και των προτάσεων που έχουν γίνει στην έκθεση του Κοινοβουλίου. Καλύπτουν τις εξής, ε, τους εξής τομείς ε, ε, υγεία και συμμετοχή, καταπολέμηση του ντόπινγκ, στατιστική, βιώσιμη ανάπτυξη, εκπαίδευση και κατάρτιση διάφορες ε, πρωτοβουλίες θα εκτελεστούν στα πλαίσια του σχεδίου δράσης ε, εμπειρογνωμόνων και βάσει και των προτάσεων ε, του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει διάφορες δράσεις, όπως για παράδειγμα έρευνες για Ό,τι αφορά συγκεκριμένα η έραση ερασιτεχνικών ε, δραστηριοτήτων, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές πτυχές ε, για τις μεταφορές ε, παικτών και σε ό,τι αφορά το σχετικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διοργανώνουμε συνόδους για στατιστικά στοιχεία και για τους αθλητικούς παράγοντες και επιπλέον έχει ξεκινήσει ένα τρίτο έτος ε, δράσεων κατά της βίας, κατά του ρατσισμού και κατά των διακρίσεων στον αθλητισμό και για να προωθηθεί η καλή διακυβέρνηση σε αθλητικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά δεν θα ολοκληρωθούν αν δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε πολυετή χρηματοδότηση. Και σωστά το Κοινοβούλιο ζητάει να προταθεί ένα φιλόδοξο προπολογισμό για τον αθλητισμό στα πλαίσια του μελλοντικού χρηματοοικονομικού πλαισίου. Χάρη στην υποστήριξή σα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πρόγραμμα πλέον, το Erasmus for All, να συμπεριλάβει ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον αθλητισμό. Το νέο πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην, ε, στους στόχους για το 2020 ως οικονομικός ε, τομέας θεωρείται ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει από μόνος του σημαντικό ρόλο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρο. Πρόεδρε. Ευχαριστώ εγώ Επίτροπε. Και τώρα να σας πω ότι θα είμαι πάρα πολύ αυστηρό σε σχέση με το χρόνο Θα σας κλείνουν τα μικρόφωνα. Αν δεν τρίτε το χρόνο σας. Έχουμε 25 ομιλητέ και μετά τη διαδικασία Catch the Eye και μετά έχουμε και τι ομιλίε ενό λεπτού. Σα παρακαλώ να δείξετε επιταρχία. Ο κ. Πάλτς για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση. Με την γνωμοδότησή μου από την Επιτροπή Οικονομικών και Μεσμαντικών Υποθέσεων, αυτό που τονίζουμε είναι ότι πέρα από την ε, διάσταση της υγείας υπάρχει και μια διάσταση οικονομικής στον αθλητισμό. Και είμαι βέβαιος ότι στον τομέα αυτό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα δημιουργηθεί κάποια υπεραξία παραπάνω. Και επί της ουσίας θα ήθελα να συνεχίσει να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας ε, στον αθλητισμό. Θα πρέπει ο αθλητισμός να παραμείνει κοντά στον πολίτη. Και αυτό είναι καλύτερο να γίνεται σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να περιοριστεί στα ζητήματα εκείνα που είναι απολύτω απαραίτητο σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το νομοθετικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τι δημόσιε προμήθειε, τον ανταγωνισμό, τα δικαιώματα διαφήμιση και το Καλώ ορίζω λοιπόν το γεγονό ότι όλα αυτά αποτυπώνονται στην έκθεση του εισηγητή και υποστηρίζω πλήρω το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και που τηρήσατε το όριο που σας ε, ε, έδωσα. Δεν βλέπω την κυρία Κόνη πουθενά. Άρα, η κυρία Κορχόλα έχει το λόγο. Αλλά ούτε και αυτή τη βλέπω. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Μάντες. Παρακαλώ ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μιλήσω τρία λεπτά. Δηλαδή, γιατί μια και έλειπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και είναι πολύ κρίμα που μια τροπολογία της Επιτροπής Δικαιοσύνης και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς για το διάλογο που ζητείται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους επαγγελματικούς οργανισμούς αθλητισμούς δεν πέρασε τελικά. Δηλαδή τι, αρνούμαστε ότι θα πρέπει να τηρούν αυτοί οι οργανισμοί ε, την οικονομική, το οικονομικό πλαίσιο, την οικονομική νομοθεσία. Ότι δεν υπάρχει τέτοια ισότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και με την ελάχιστη διάρκεια των συμβάσεων, ότι υπάρχουν προβλήματα με την αντιμετώπιση των επαγγελματιών στον τομέα του αθλητισμού, ότι υπάρχουν γενικά προβλήματα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει διάλογο με τους επαγγελματικούς, ε, ε, με οργανισμούς επαγγελματιών για να είμαστε βέβαιοι ότι και η νεολαία θα μάθει από αυτά, αυτές τις ρυθμίσεις. Ε, θα ήθελα να συμφωνήσω λοιπόν με όλα αυτά που έγραψε ο συναδελφός Βίζας, αλλά κρίμα που δεν ελήφθησαν υπόψη όλα αυτά από την Επιτροπή ε, Ευχαριστώ κύριε Μποσκούρτ. Κυρία Εμινέ Μποσκούρτ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, ο αθλητισμός αποτελεί ε, πολύ σημαντικό για εκατομμύρια Ευρωπαίους. Ε, και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει μια καλή πολιτική για τον αθλητισμό και να διορθώσει τα σφάλματα. δυστυχώς φαίνεται ότι οι καλές προθέσεις δεν ε, συνοδεύονται από αναλογές πράξεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Το 2010, 1.100 ε, ανήλικοι αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμβάσεων σε επαγγελματικά ε, συμβόλαια ως εξαίρεση. Και, για παράδειγμα, οι πράκτορες θα πρέπει να έχουν ένα κώδικα διοντολογίας, μια μαύρη λίστα, να τους επιβάλλονται κυρώσεις γιατί η Ευρώπη αντιμετωπίζει διάφορα ατυχή περιστατικά σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πάρει αυτά στα σοβαρά, να εφαρμόσει νομοθεσία που θα απαγορεύει διακρίσεις, να διεξάγει σχετικές ε, εκστρατείες για να καταστήσει σαφές ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διάκριση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε εποχές ε, λαϊκισμού και εξτρεμισμού γιατί οι εγκληματίες είτε μέσα στο γήπεδο είτε έξω από το γήπεδο επηρεάζουν και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να λαμβάνονται δράσεις από όλα τα κράτη και η Ευρώπη και οι αθλητικές οργανώσεις θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να συνεργαστούν με την Europol και την Eurojust. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον αθλητισμό. Αυτό το χρειαζόμαστε κατεπηγόντως. Προς το παρόν είναι υπερβολικά ε, μη δεσμευτικέ αυτές οι αρχές που έχουν τεθεί. Φυσικά το fair play αποτελεί το στόχο μας, αλλά αυτό, όλα αυτά χρειάζονται μια ισχυρή πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σενίσιν για ένα λεπτό. Αλλά δεν τη βλέπω στην αίθουσα, οπότε συνεχίζουμε με τον κύριο Σκούρια. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, εισηγητή Φίσας για την εξαιρετική του δουλειά. Είναι για μια, έκανε μια έκθεση την οποία θα χαρακτήριζα πλήρη και η οποία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον τομέα του αθλητισμού. Δούλεψε πάρα πολύ καλά και με τους σκιώδεις ε, συνεισηγητές του. Και θέλω φυσικά να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επίτροπο Βασιλείου. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μήνυμα αυτό που στέλνει η συγκεκριμένη έκθεση. Ιδιαίτερα μια Ολυμπιακή χρονιά που είναι θα έλεγα το πιο σημαντικό σημείο του αθλητισμού στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη την κοινωνικοποίηση που προσφέρει ο αθλητισμός. Είναι επίσης μέσω καταπολέμησης των διακρίσεων. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιες γυναίκες να αθληθούν σε χώρες όπως το Ιράν. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσα Αθλητισμού στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας η οποία γίνεται ανάμεσα στις λεγόμενες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το θέμα της καταπολέμησης φυσικά του τζόγου, επίσης το ντόπινγκ είναι κάτι το οποίο σημειώνεται σωστά στην έκθεση. Έχουμε νέες αρμοδιότητες, τις οποίες μας έχει δώσει άλλωστε η συνθήκη της, της Λισαβόνας στον συγκεκριμένο τομέα. Ιβάννα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την συνενετική του στάση. Συζητήσαμε το σύνολο του κειμένου του αναλυτικά και μπορέσαμε να βρούμε αρκετές κοινές θέσεις, ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο πέτυχε ο κύριος Φίσας έχει σημασία. Λόγω ακριβώς της σημασίας που έχει ο αθλητισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατετέθησαν εκατοντάδες τροπολογίες. Και για μια ακόμη φορά θέλω να συγχαρώ για αυτό τον εισηγητή. Η προσπάθειά του δεν είναι απλά μια περιγραφή της ισχύουσας κατάστασης στον τομέα του αθλητισμού σήμερα δεν περιορίστηκε ο κύριος Φίσας σε μια απλή παρουσίαση της κατάστασης. Αντίθετα, η έκθεση περιλαμβάνει τολμηρές ιδέες, τολμηρές πρωτοβουλίες και έχει σημασία να ακολουθήσουμε τις προτάσεις της τολμηρές, σαν παράδειγμα το καθεστώς των ανηλίκων παιδιών, που εμπλέκονται σε αθλητικές δραστηριότητες, το θέμα του στοιχηματισμού στον αθλητισμό κτλ. Ξέρουμε ότι το σπορ δεν είναι απλά ε, μια διασκέδαση. Είναι κάτι που έχει σημασία και για τη δημόσια υγεία και για την παιδεία και για την μη βία και για την οικονομία επίσης όπως και για άλλους τομείς. Ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει και να συνεισφέρει σε μια σωστή και με καλές επιδόσεις οικονομία. Μόνο το 1% του συνολικού προϋπολογισμού του Εράσμους αφιερώνεται στα αθλητικά. Αυτό δεν είναι επαρκές. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες πιστώσεις στον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Aylward, φιλελεύθερη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια σωστή αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Έχει προκαλέσει πάρα πολύ ενδιαφέρον η έκθεση αυτή και από αθλητές και από εθελοντές και από αθλητικές ομάδες και οργανώσεις και συλλόγους. Ενώνει ο αθλητισμός και πλουτίζει τη ζωή μας. Μια ευρωπαϊκή πολιτική στον αθλητισμό δεν είναι θέμα εναρμονισμού. και δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει οι αρμόδιες ενώσεις ε, των σωματείων ε, και των αθλητών κάθε χώρας να είναι υπεύθυνε για τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουν στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της αντιμετώπισης του ντόπινγκ, ε, θέματα τα οποία δεν μπορεί να αποκρυβούν. Νομίζω ότι έτσι θα δημιουργήσουμε μια σωστή αθλητική πολιτική χωρίς αποκλεισμούς. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα η οποία ε, ε, έχει την πιο παλαιά θα έλεγα ερασιτεχνική αθλητική ένωση, την Ένωση ε, Κελτικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων, ένα εκατομμύριο μέλη, ο ρόλος των εθελοντών και των ερασιτεχνών είναι πάρα πολύ σημαντικός για κάθε κοινωνία και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό για τα ερασιτεχνικά αθλήματα. Βοηθά λοιπόν ο αθλητισμός την οργάνωση της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο παράγει καλό για την κοινωνία και θα πρέπει επίσης εδώ να δούμε και τι γίνεται με τον ρόλο των δημοσιογράφων όταν αναφέρονται σε αθλητικές διοργανώσεις. Το κοινό διψά και έχει ανάγκη από σωστή και αντικειμενική ενημέρωση. Ευχαριστώ το λόγο. Έχει κυρία Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, Θέλω ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Φίσας για την έκθεσή του και τους και τους ηγητές ε, για τη συμβολή τους. Η πολιτική ομάδα μας είναι υπέρ της ε, ευρωπαϊκής δράσης ε, στον τομέα του αθλητισμού, όπω αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαστε υπέρ και των προτάσεων του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι η έκθεση ε, μιλάει για την υποστήριξη παραδοσιακών σπορ και παιχνιδιών ως τμήματων σημαντικών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κάποια παραδοσιακά παιχνίδια και παραδοσιακές μορφές αθλητισμού ε, κινδυνεύουν να αφανιστούν. Θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε λοιπόν. Επίσης μας ενδιαφέρουν κάποιες κοινωνικές πτυχές των επαγγελματιών αθλητών και αθλητριών. Μερικές φορές το μέλλον τους είναι αβέβαιο όταν τερματίζεται η αθλητική τους σταδιοδρομία. Το θέμα αυτό υπογραμμίστηκε και από το συνδικά Συνδικάτο Αθλητισμού και Τουρισμού στη συζήτηση που έγινε για το θέμα αυτό. Η Ευρώπη θα πρέπει να προωθήσει το κοινωνικό της μοντέλο και να βοηθήσει τις, τους κοινωνικούς όρους διαβίωσης ε, της ιδιαίτερης αυτής κατηγορίας εργαζομένων που είναι οι επαγγελματίες αθλητές. Έκλεισε λοιπόν προς τα κράτη-μέλη να βρεθούν τρόποι για να ελαφρυνθεί το οικονομικό βάρος για τους αθλητές ιδιαίτερα που δεν αμείβονται με υψηλέ αμοιβέ. Επίσης χρειαζόμαστε έναν κοινό ορισμό του όρου των ε, συνταξιούχων ε, αθλητών και προπονητών. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο κοινό ορισμό. Η γνωμοδότηση τη Νομική Επιτροπή περιλαμβάνει έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με, όλους, με όλε τι επαγγελματικέ ε, αθλητικέ οργανώσει για να αντιμετωπιστούν ε, τα προβλήματα που οφείλονται στι διαφορές, ε, νομικέ διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών για τα συμβόλαια του. Ευχαριστώ για δύο λεπτά, κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ σημαντική η θέση του αθλητισμού στην Ευρώπη. Όχι μόνο παράγει εκατομμύρια ευρώ και πολλέ θέσει εργασία, αλλά δίνει μεγάλη χαρά σε πολλού. Και εγώ είμαι μεταξύ αυτών με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ε, θα έπρεπε να είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ερευνήσει τρόπου ε, για, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό και την ε, αθλητισμό. Αυτή η έκθεση αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία γιατί στρέφεται στο πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το πόσο δημοφιλή είναι κάποια αθλήματα και τι μπορεί να κάνει το αθλητισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το αντίστροφο. Επικεντρώνεται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν λαμβάνει υπόψη, για παράδειγμα, αεραστεχνικές οργανώσεις όπως θα έπρεπε. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάσει ε, πράγματα όπως η καταπολέμηση του ντόπινγκ και το καθεξής. Αλλά η έκθεση πάει υπερβολικά μακριά. Γιατί καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει συλλογικά και όχι τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση. Επίσης ε, προτείνει ειδικό καθεστώς φόρων και ε, άπτεται θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία όλα αυτά τα θέματα είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών και το πιο επιζήμιο είναι που προτείνει να υπάρχει ευρωπαϊκή σημαία και όχι εθνική σημαία στις ε, ευρωπαϊκές ομάδες. Και η πρόταση αυτή είναι εξωφρονική και περιττή. Ο αθλητισμός έχει πολύ ιδιαίτερη θέση στον Ηνωμένο Βασίλειο και οι εθνικές μας ομάδες αποτελούν τμήμα της εθνικής μας κληρονομιάς και ταυτότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιβάλλει την ταυτότητά της ε, και αυτό δεν προάγει τον αθλητισμό, προσπαθεί μόνο να προσθέσει αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να υπερψηφίσω αυτή την έκθεση αύριο. Ευχαριστώ. Βλέπω πίσω σας μια πράσινη γαλάζια κάρτα. Δέχεστε την ερώτηση κυρία Μακλάρκιν. Καλώς έχει το λόγο. ως προέθλητης και σπόνσορ του, ε, της γυναικής ομάδας του Cambridge, του Πανεπιστήμιου του Cambridge, θα έλεγα ότι μαντεύονται σε 15-20 χρόνια θα φοράν μπροστά στο, στο προστινό μέρος, στο πίσω μέρος της ε, ε τους το σύνθημα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Μακλάρκιν, όχι. Οπότε προχωρούμε στους επόμενους ομιλητές. Η κυρία Βερζιά για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο αθλητισμός ε, ε, ε, θεωρήθηκε μόνο υπό το πρίσμα της αγωνιστικότητας και κρίθηκε ως αμυγός οικονομική ενέργεια. Επιτέλους αναγνωρίζεται και η παιδαγωγική, πολιτιστική, κοινωνική και ε, πτυχή υγείας του αθλητισμού. Επιμένει στο ρόλο των θελοντών και την ανάγκη κατάλληλου νομικού και φορολογικού πλαισίου. Χαιρόμαστε για όλες τις προτάσεις της έκθεσης αυτής. Θα πρέπει να επενδύσουμε και στο μαζικό αθλητισμό. Επίσης, σωστή διάκριση μεταξύ του επαγγελματικού και του αεραστεχνικού αθλητισμού. Είναι σημαντικά τα, κρατικά ενδύλια και να έχουμε ίση πρόσβαση χωρί. Διακρίσει διακρίσεις στον αθλητισμό. Χρειαζόμαστε επίσης ε, πραγματική εταιρική σχέση με τις αθλητικές ομοσπονδίες. Τα κράτη θα ε, διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να εφαρμοστεί το ήθος ε, του αθλητισμού και μια συγκεκριμένη διοντολογία και στον ερασιτεχνικό και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Βέβαια, τι, γίνεται, τι κάνουν οι μυστικές αρχές ό,τι αφορά τα έκτροπα που παρατηρούμε πολλές φορές στον αθλητισμό. Υποβάλαμε μια πρόταση ε, σε ό,τι αφορά το μονοπόλιο των ε, χωρών. Ε, είχαμε την σχετική νομολογία του ΔΕΚ, δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας. Είπαμε να θέλουμε τα κράτη-μέρη να εξασφαλίσουν τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των αθλητών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και το δικαίωμα για επαγγελματική ανακύκλωση. Αλλά δεν αρκούν τα ωραία λόγια. Χρειαζόμαστε έργα και το πρίσμα της εσωτερικής ε, αγοράς και του ανταγωνισμού θα πρέπει να τεθεί στη σωστή διάσταση, να αναγνωριστούν οι αθλητές και η αξία του αθλητισμού ως σημαντικό εργαλείο προσωπικής ε, και συλλογικής αυτοεκπλήρωσης. Ευχαριστώ κύριο Σινότχαλ. Mr. President, e flag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 Ποτέ δεν ήταν τόσο λίγο δημοφιλής η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά με τη ματαιοδοξία σας θέλετε να φαίνονται τα αστέρια σας. Λέγεται σε μία απόφαση της FIFA ότι η ομάδα η οποία μεταφέρει πολιτικά σήματα ή πολιτικά συνθήματα θα υποστεί κυρώσεις από τη FIFA. Πώς λοιπόν πιστεύετε ότι έχετε δικαίωμα να παρεμβαίνετε και να ζητάτε από χώρες να παραβιάσουν τον νόμο. Αυτό είναι υποκριτικό. Η Πολιτική Ένωση είναι μια πολιτική οργάνωση. Λέτε στην παράγραφο 20 ότι η πολιτική προπαγάνδα θα πρέπει να απαγορευτεί. Αυτό είναι υποκριτικό. Οι αθλητές φορούν την εθνική τους φανέλα και όχι φυσικά τη φανέλα της Ένωσης, προφανώς. Βλέπω μπλε κάρτα Παρακαλώ. Τώρα ψήμετε οτάσκου. Κύριε Νάτχολ, δέχεστε την ερώτηση από τον συνάδελφο. Κύριε Νάταλ, συμφωνώ μαζί σα, αλλά δεν νομίζω ότι πάτε αρκετά μακριά, γιατί αυτό σίγουρα είναι ντροπιαστικό και προφανώ ε, εξοργίζει του οπαδού. γιατί για παράδειγμα στο παγκόσμιο κύπελο αν ε, προτάσσεται η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Ομάδα, ποιον υποστηρίζει ο παδός, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την ομάδα του. Δεν είναι το ίδιο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καν χώρα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι χώρα. Και αυτό που προσπαθείτε να ε, δημιουργήσετε είναι επικίνδυνο, γιατί όπως και η Σιωβετική Ένωση, ε, οι ομάδες χωρών αυτές σπάνε είτε με ειρηνικό τρόπο, όπω η Τσεχοβεσλοβακία, που ελπίζω να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, ή με αιματηρές ε, επαναστάσει, το οποίο και φοβάμαι ιδιαίτερω. Ε, Ευχαριστώ το συγγνώμη. Στον ομιλητή έχετε ήδη ζητήσει ε, μπλε κάρτα και δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να προχωρήσουμε. Ε, κυρία για λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση για την Ευρωπαϊκή Διάσταση του Αθλητισμού είναι πάρα πολύ σημαντική. Το άρθρο 156 ε, καλύπτει την ε, ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για θέματα τέτοια. Σκοπός μας είναι η προώθηση της υγείας Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε στην χώρα μου και στην περιφερειά μου, το Ζάλτσμπουργκ. Εμείς έχουμε πολλές ε, χειμερινές ε, ε, εκδηλώσεις και πολλά χειμερινά αθλήματα και αυτό, σε αυτά θα συμμετέχουν όλες οι οικογένειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αθλητισμός και για τους πρεσβύτερους της κοινωνίας και θέλουμε να συμμετέχουν και πιο πολλές γυναίκες στην διαδικασία ε, σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις τις αθλητικές, σε ό,τι αφορά τον ντόπινγκ και την διαφθορά στον ε, αθλητισμό, ελπίζουμε να αναφερθούν μόνο αυτή τη φορά και να βελτιωθούν στο μέλλον και να μην χρειαστεί να ξαναναφερθούν. Να ευχαριστήσω πάλι τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενος ο είναι η κυρία Ματέρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πεπισμένος ότι ο αθλητισμός έχει έναν βασικό εκπαιδευτικό ρόλο, παιδαγωγικό ρόλο, πολιτιστικό ρόλο. Ο αθλητισμός είναι ταυτόχρονα ένα μέσο ενσωμάτωσης, αντιπαράθεσης, σύγκρισης και ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να δώσουμε μια μεγαλύτερη ομοιογένεια και ταυτόχρονα να καταστήσουμε τον αθλητισμό ελκυστικό και παραγωγικό χωρίς διακρίσεις για όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να τον περιορίσουμε στο εσωτερικό ενός κράτους γιατί ενδιαφέρει το σύνολο των μελών ε, της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβει γιατί ε, θα έλεγα διατρέχει μια οξία και συνεχή κρίση λόγω εγκληματικών δραστηριοτήτων Αναφέρομαι σε σκάνδαλα με απαγορευμένες ουσίες ή επίσης και τα στοιχήματα και τα λοιπά και τα φτιαγμένα παιχνίδια, τα στημένα συγγνώμη παιχνίδια. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει ένας μεγαλύτερος έλεγχος από πλευράς των ευρωπαϊκών οργάνων στον τομέα του σπορ, έτσι ώστε να αποτρέψουμε τις παρεκκλήσεις οι οποίες σημειώνονται μια λεπτομερής και εφαρμόσιμη περιγραφή θα επιτρέψει, θα έλεγα, τα επίπεδα της, θα βελτιώσει τα επίπεδα της αθλητικής διακυβέρνησης. Είναι απαραίτητο να παρέμβουμε για να ρυθμίσουμε επίσης και τις δραστηριότητες των μάνατζερ, τις μεταγραφές, την καταπολέμηση των απατών, την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και άλλων χημικών. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Childers. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απογευματινή συζήτηση, η βραδινή συζήτηση μάλιστα, μάλλον, έδωσε επιχειρήματα στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει πιο αποτελεσματικά τον αθλητισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ 25 ε, χρόνια εργάστηκα ως επαγγελματία ε, σε θέματα πνευματικής και ψυχικής υγείας. Δεν έχει ε, αναγνωριστεί υπέρ της, ο ρόλος του αθλητισμού για την ψυχική υγεία, γιατί δημιουργεί, προκαλεί έκρηση ενδοκριν, ενδορφινών και βελτιώνει την ψυχική κατάσταση και την ευεξία. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη και αυτό ο ρόλο του αθλητισμού και περιμένω πρόοδο στον τομέα αυτό. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Τάκουλα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ε, συγχαρώ για την εκλογή σας ως αντιπρόεδρος και να σας συγχαρώ και για τη συζήτηση που διεξάγουμε εδώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Βίσας για την ε, πολύ καλή του έκθεση και θα ήθελα να πω ότι η Επίτροπος έχει εργαστεί πολύ αποτελεσματικά υπέρ του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ο αθλητισμός αποτελεί το μεγαλύτερο κίνημα πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα θα έπρεπε να διαδραματίζει σαφή ρόλο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει έρθει λοιπόν η στιγμή να περάσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Η έκθεση αυτή δεν είναι μια καλή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτά που είναι απαραίτητα ο αθλητισμός έχει θετικές ε, ε, συνέπειες για την υγεία, αλλά δράει και με συλλογικό τρόπο για την ε, κοινωνική αλληλεγγύη. Και γι' αυτό είναι πολύ, μάλλον είναι πολύ σημαντικός ο αθλητισμός και για την καταπολέμηση του ρατσισμού στην Ευρώπη. Φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα θέματα χρηματοδότησης και θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ότι στον προϋπολογισμό θα πρέπει να βρούμε επαρκείς πόρους για τον αθλητισμό προκειμένου να αποτρέψουμε και να ξεπεράσουμε και τα εθνικά μονοπόλια σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των επιθυμητών μέτρων. Και τέλος να πω δύο λόγια για το θέμα της ε, σημαία. Στην Ευρώπη επικρατούν διάφορες ευρωπαϊκές ε, σημαίες. Εγώ θεωρώ ότι αν υποστηρίζει κανείς την ομάδα που υποστηρίζει την ομάδα του στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα όταν παίζουν οι Άγγλοι, θεωρώ ότι αυτό θα έδινε, μάλλον μια ευρωπαϊκή σημεία θα έδινε μια νέα πτυχή. Κύριε Γιανακουδάκη, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να, χαρώ, να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε για την εκλογή σας. Ως Βρετανίδα ανταλαμβάνομαι το σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στη ζωή μας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, επεβαίνει σε θέματα αθλητισμού. Θα πρέπει να επικεντρωθεί σε θέματα ανάπτυξη, απασχόληση και ενιαία αγορά. Γιατί χώνατε και στον αθλητισμό. Η έκθεση αυτή πέρασε από 7 επιτροπέ και ήμουν σκιώδη συγγήτρια τη ομάδα μου σε δύο από αυτέ. Ε, είχα την πρόθεση να μιλήσω σήμερα για τις Βρετανίδες που είναι ε, Όπω η Ρεμπέκα Άντεκτον, η Κέλλη Χόμς και η Πόλα Ράτκλιφ, ηρωίδε αθλήτριε, για εκατομμύρια ε, συμπολίτε τους. Ε, στην εκλογική μου περιφέρεια του Λονδίνου με χαρά θα, θα υποδεχθούμε τους ε, συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς. Δεν μπορώ όμως να μιλήσω για αυτά γιατί θέλω να καταγγείλω την ε, πρόταση της έκθεσης να χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή σημαία στις αθλητικές εκδηλώσεις και να περιλαμβάνεται και στο, στην ένδυση των αθλητών. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ξοδεύουμε σε εποχές λιτότητας κονδύλια για να συμπεριληφθεί η ευρωπαϊκή σημαία σε αθλητικές εκδηλώσεις. Θα πρέπει η φυσαλίδα των Βρυξελών να θυμάται ότι διανύουμε χαλεπούς καιρούς. Σας ευχαριστώ. Γαλάζια κάρτα Έχετε, δέχεστε την ερώτηση, κυρία Γιανακουδάκη. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω την ομιλητηρία σε ό,τι αφορά το σχόλιο της για την Ευρωπαϊκή Σημαία. Αναφέρεται στην έκθεση ότι θα πρέπει να είναι τελείως προαιρετικό και να αναπόκειται στα κράτη-μέλη η συμπερίληψη της Ευρωπαϊκής Σημαίας. Το απολύτως προαιρετικό πώς το καταλαβαίνει, γιατί, γιατί επέμεινε, πώς το ερμηνεύει το τελείως προαιρετικό. Ναι, πολύ ευχαρίστω να σας πω. Τελείως προαιρετικό. Δεν θα πρέπει καν να αναφέρεται σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το στάδιο. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τον αθλητισμό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να στηρίξουμε τον αθλητισμό. Να υποστηρίξουμε τις εθνικές μας ομάδες. Δεν νομίζω ότι στην έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται κάτι τέτοιο προαιρετικά ή ε, αλλιώς. Η έκθεση θα ήταν καλύτερη αν δεν είχε αυτό το προαιρετικό, ε, αν δεν, είχε τίποτα, αν δεν αναφέρεται τίποτα για το θέμα αυτό. Συνεχίζουμε, κύριε Ζουμπέρ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε θεωρούμε θεμελιώδες για την προσωπική κοινωνική ανάπτυξη, την οικουμενική και δωρεάν πρόσβαση στον αθλητισμό με ποιότητα. Και θα πρέπει αυτό να εξασφαλίζεται σε όλους χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τα κράτη-μέλη με υποστήριξη των ε, αθλητικών οργανώσεων αλλά και μέσω των σχολείων γιατί και τα σχολεία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πραγωγή του αθλητισμού. Η έκθεση ακολουθεί σωστή κατεύθυνση ό,τι αφορά την πρόθεση του αθλητισμού. Προτείνουμε συγκεκριμένο προπολογισμό και φιλόδοξο για την πολιτική αθλητισμού. Ε, ε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τον αριστεχνικό αθλητισμό και τα τεράστια έσοδα από τα στοιχήματα. Αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Θεωρούμε ότι τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, κατά και αποδυναμώνουν το, κράτος, το κοινωνικό κράτος και τη δημόσια, ε, το δημόσιο σχολείο, η νέα αυτή πολιτική δεν συνάδει καθόλου με τις προτάσεις της έκθεσης. Σας ευχαριστώ για δύο λεπτά, κύριος Μπόρης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, θερμά τον ε, κύριο Φίσας που για ένα χρόνο και ασχολήθηκε με την πολύ σημαντική αυτή έκθεση. Είναι ε, μια έκθεση που μιλά για τη νέα πολιτική ε, αθλητισμού που μπορεί να αποκτήσει τελείω διαφορετικό χαρακτήρα μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Έχουμε ε, χιλιάδε οργανώσει και αθλητέ που περιμένουν ε, αποτελέσματα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ θερμά τον κύριο Φίσα. Πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική αθλητισμού τα επόμενα χρόνια. Θα εξαρτηθεί από εμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και από εσά, κύριε Επίτροπε, γιατί έχουμε πολύ σημαντικές συστάσεις στην έκθεση και ελπίζω να εφαρμοστούν και εμπράκτο οι σημαντικές αυτές συστάσεις. Και η διασφάλιση αυτών των τριών στοιχείων του οικονομικού στοιχείου, του πολιτιστικού ε, ε, στοιχείου του αθλητισμού είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι μπορούμε επιτέλους να εφαρμόσουμε και αποτελεσματικά την πολιτική αθλητισμού. Θα πρέπει να δούμε τον κανονισμό για τους μάνατζερ, για τη διαφάνεια του συστήματος, ε, θα πρέπει να αναδείξουμε τα νέα ταλέντα και όχι να τα εκμεταλλευτούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές σχετικές προτάσεις ε, του κυρίου Φίσας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το επάγγελμα του, του εκπροσώπου του αθλητή, του μάνατζερ. Επίσης, η χρηματοδότηση του fair play. Είναι πολύ σημαντικό το fair play, το εφαγωνίζεστε και θα πρέπει να προωθηθεί ήδη από το σχολείο, γιατί έχουμε και το παθολογικό φαινόμενο του στήσιματος των αγώνων. Πολύ συχνά το στήσιμο των αγώνων έχει και μαφιόζικο χαρακτήρα. Υπάρχει και το θέμα του αθλητικού τουρισμού. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας, ε, κύριε Επίτροπε. Ε, θα μπορούσαμε διαρθρωτικά κονδύλια και κυρίως ε, κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου να τα αφιερώσουμε στη βελτίωση της βάσης του αθλητισμού για να προωθήσουμε τον αθλητισμό και τον, αεραστεχνισμό και, τον και τον επαγγελματικό. Θα ήθελα να επενέσω τον εισηγητή γιατί είναι εξαιρετικό και ελπίζω να γίνει δεκτό και από τα κράτη-μέλη στην πολύ σημαντική χρονιά και του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, ε, και του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και των Ολυμπιακών Αγώνων. Η κυρία Σιμόλκοβα. Ε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να, υποστηρίξω. Σε ό,τι αφορά τα... ότι θα πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία αρκετέ αθλητικέ εγκαταστάσει, γιατί πάνω απ' όλα ο αθλητισμό μπορεί να ενισχύσει την υγεία και ο αθλητισμός θα πρέπει να ενσωματώσει και του κοινωνικά αποκλεισμένου. και παράλληλα να καταπολεμήσει κάθε διάκριση. Ο αθλητισμό μπορεί να ωφελήσει όλες τις γενιές σε ό,τι αφορά την υγεία, την κοινωνική διάσταση, την πολιτισμό ή την οικονομία για την νεολαία. Ο αθλητισμός αποτελεί ένα μέσο για τον ελεύθερο χρόνο τους και κατά την καταπολέμηση για παράδειγμα της χρήσης ναρκωτικών. Ως γυναίκα θα ήθελα να υπάρχει πιο πολύ υποστήριξη για τις γυναίκες αθλήτερες και να υπήρχε πιο πολύ ισότητα ευκαιριών στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Κέλλη για δύο λεπτά. Ε, ε, ε, Καταρχά να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για την τραγωδία στην Αίγυπτο Χαίρομαι κατά τα άλλα που παίρνω μέρος στη συνάντηση αυτή και στη συζήτηση αυτή γιατί τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκα πολύ με τον αθλητισμό. Ήμουν πρόεδρος της ε, Ομοσπονδίας Κελτικού Αθλητισμού. Νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα με την έκθεση αυτή και σε σχέση με αυτά τα οποία προβλέπει η Λισαβόνα να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες, ελπίζω να γίνουν δεκτές, ιδιαίτερα για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, σχετικά και με τη γραπτή δήλωση που υιοθετήθηκε πέρυσι. Επίσης να υπάρξουν μέτρα και για τον αθλητισμό τουρισμό, για τα διαφορετικά ταμεία που θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ιδιαίτερα τις παραδοσιακές αθλητικές δραστηριότητες που είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες αλλά χρήζουν βοήθεια όπως στη χώρα μου. Ένα επίσης επιχείρημα που μπορούμε να προτείνουμε είναι ότι ο αθλητισμός άμεσα ή έμεσα εμπλέκει 50 εκατομμύρια ανθρώπους και ταυτόχρονα διασφαλίζει το 3,6 του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. σχετικά με την πρόταση την εθελοντική για τη χρήση της Ευρωπαϊκής Σημαίας ε, δεν μου κάνει κάποια αρνητική εντύπωση. Μπορούμε κάλλιστα να τη χρησιμοποιούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του αθλητισμού είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό και επίσης να επιμείνουμε και για την αύξηση του προϋπολογισμού του έρασμος για τις αθλητικές δραστηριότητες, ανταλλαγές. Ευχαριστώ κύριος Μπέλετ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, καλησπέρα και συγχαίρω τον συνάδελφο Σαντιάκο Φίσας για την εξαιρετική αυτή έκθεση που μας παρουσίασε. Ο αθλητισμός από ε, κοινωνικής άποψης ε, έχει τόσα πολλά πλεονεκτήματα που δεν χρειάζεται καν να τα αναφέρουμε. Ωστόσο πρέπει να τα τονίσουμε. Είναι σημαντικό να αφήσουμε χώρο για μέσα που θα εξασφαλίσουν ε, την καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών στον αθλητισμό. Και γι' αυτό, Πρόεδρε και αξιότιμη Επίτροπε, θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα προς τους Βρετανούς ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι έχουν φύγει βέβαια ήδη, να δείτε τι συνέβη σήμερα στην Αίγυπτο, όπου χάθηκαν οι ζωές ε, δεκάδων οπαδών να δούμε τι συνέβη στη Βιέννη σήμερα, όπου καταδικάστηκαν ε, δεκάδες οπαδοί λόγω χρήσης βίας σε γήπεδα και γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή πολιτική και θα αναφέρω αυτά που λέει η έκθεση του κυρίου Φίσας απαγόρευση εισόδου σε γήπεδα όλων των, όλων των χούλιγκαν και αυτό θα πρέπει να ισχύει και σε διεθνείς αγώνες. Αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον αθλητισμό. Γι' αυτό θα σας υποστηρίξουμε, Επίτροπε, μια βάση δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών για χούλιγκαν που χρησιμοποιούν βία και είναι ρατσιστέ. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπω είπαν οι συνάδελφοι, η καταπολέμηση του ντόπινγκ, η καταπολέμηση α, ε, των, της Γι' αυτό λοιπόν, συνάδελφοι, σε αυτά θα πρέπει να επικεντρωθούν παρά να κάτσουμε να γκρινιάζουμε όλο το βράδυ για την Ευρωπαϊκή Σημαία που θα εκτυπωθεί ή όχι σε μια μπλούζα. Και το υποστηρίζω άλλωστε απόλυτα. Όπω είπε ο συνάδελφο Κέλλη, 100% σε θελούσια βάση θα γινόταν κάτι τέτοιο, με 100% σεβασμό τη ε, επικουρικότητα. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Και τώρα η διαδικασία κάτσε Έχουμε πολλούς ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα πρέπει να περιορίσουμε τον αριθμό των ομιλητών με τη σειρά που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κ. Νικολάσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ο αθλητισμός αποτελεί μία από τις λίγες δραστηριότητε που ε, καταργεί τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων χωρίς να λαμβάνει δηλαδή υπόψη ε, θέματα θρησκείας, ε, κοινωνικού στάτους και συμβάλλει επίσης σε έναν υγιή τρόπο διαβίωσης. Ενισχύει την υγεία του Ευρωπαίου πολίτη ο αθλητισμός. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίζουμε πιο πολύ τους ε, αθλητές. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και σε πολιτικό επίπεδο για τους πολίτες. Ο αθλητισμός αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία με την οποία δημιουργείται μια αισιόδοξη αντιμετώπιση της κοινωνίας. Επίσης, ο αθλητισμός έχει και εκπαιδευτικέ ε, ιδιότητες, γιατί αναπτύσσει το άτομο στα πλαίσια του εφαγωνίζεστε. Γι' αυτό, λοιπόν, υποστηρίζουμε τόσο πολύ τον αθλητισμό και θεωρούμε ότι η έκθεση περιλαμβάνει πάρα πολύ καλές ιδέες. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα για ένα λεπτό. Κυρία Τσικάου, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού θα ήθελα να πω ότι οι αθλητικές εκδηλώσεις συμβάλλουν και στην ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποιες συνέργειες μεταξύ τουρισμού και αθλητισμού, εξυγχρονίζοντας ε, τις υποδομές. Ένα παράδειγμα συνέργειας μεταξύ τουρισμού, μεταφορών και αθλητισμού είναι το τουριστικό δυναμικό του, της ποδηλασίας. Έχουμε 14, 14 μονοπάτια ποδηλατικά, 70.000 χιλιόμετρα ανά την Ευρώπη. Αυτό προωθεί την κοινωνική ένταξη, ε, την ανάπτυξη του τουρισμού και τη προστατεύει και το περιβάλλον. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τέτοιους ποδηλατοδρόμους διασυνοριακούς και ε, γιατί όχι τους ποδηλατοδρόμους που θα περνάνε ε, από θα, θα, θα περνάνε κατά μήκος του Δούναβη. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε ε, κάποια προγράμματα κινητικότητα των πολιτών και να ενισχύσουμε τις υποδομές που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή αθλητικών οργανώσεων. Ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό. Είναι θετικό το γεγονός ότι μέσω της συνθήκης ε, προωθούνται το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει γιατί δεν ε, ασκείται αρκετά και αυτό οδηγεί σε διάφορα προβλήματα όπως υπάρχει σαρκία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθηθεί ο αθλητισμός. Αυτό υποστηρίζει και την υγεία παράλληλα και συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος και για τα συστήματα ασφάλισης. Έτσι λοιπόν, μέσω του αθλητισμού, ε, ο αθλητισμός θα έπρεπε να αποτελεί μια βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και σε διάφορου διαγωνισμού. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, διοργάνωση των πολιτών ανά αθλητικές οργανώσεις και αυτό θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όλων. Ευχαριστώ πολύ και τώρα κυρία η Βόρεια Ιρλανδία παθιάζεται με τον αθλητισμό. τελευταίο, τον τελευταίο 1,5 χρόνο πήραμε και τρία παγκόσμια μετάλλια και αυτό είναι ασυνήθιστο για ένα τόσο μικρό τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα σχετικά με τη σημαία βέβαια δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ικανοποιήσει κανέναν και φυσικά τους οπαδούς της χώρας μου, ενώ η σημαία του Όλστερ προφανώς έχει κερδίσει τις καρδιές τους για πάντα. Λέει η έκθεση ότι οι διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις είναι ένα επίπεδο αναφοράς και θα πρέπει να μην γίνονται δεκτές ε, οι αποκτήσεις με συνοπτικούς τόπους ε, ε, ηθαγενειών για αθλητές. Είδαμε ότι στην Ιρλανδία, σαν παράδειγμα, πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίοι ε, είχαν εκπροσωπήσει τη Βόρεια Ιρλανδία σε επίπεδο εφηβικού αθλητισμού αλλά πήραν την υπηκότητα της δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σημειώσουμε. Ευχαριστώ, Επιτροπέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η Σλοβακία στην τελευταία εκλογική ε, περίοδο και ο Επιτροπός Φίγκελ ε, έθεσε μεγάλη προτεραιότητα στο θέμα του αθλητισμού. Επιτρέψτε μου παρακαλώ να αναφέρω και να παραθέσω κάτι από μια ομιλία του, ότι ο αθλητισμός αναπτύσσει ε, αρχές και αξίες που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της δημοκρατίας. Συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήματα και παράλληλα κρύβει πολλά μειονεκτήματα. προβλήματα όπως ο ρατσισμός ε, και το ντόπινγκ ε, σκοτώνουν τον αθλητισμό και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά χρειαζόμαστε κανόνες. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι είμαι θελοντική ε, πρόεδρος μιας ομάδας χόκεϊ επιπάγου και θεωρώ ότι δεν υπάρχει πραγματική ισότητα στον αθλητισμό. Ευχαριστώ κύριε Σματούλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μα για την εξαιρετική του έκθεση που είναι και πολύ επίκαιρη γιατί έχουμε μια γενική συζήτηση για το μέλλον του αθλητισμού. Ο αθλητισμός έχει τεράστιες συνέπειες ε, στην υγεία, στον τουρισμό, στην ε, κοινωνική ευημερία, στην πρόθεση της ειρήνης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως και τον ερασιτεχνικό και τον επαγγελματικό αθλητισμό. Γνωρίζουμε ότι οι επενδύσεις στον αθλητισμό σημαίνει ότι περιορίζουμε τις επενδύσεις σε θέματα δημόσιας υγείας. Μην ξεχνάμε όμως ότι και οι ηλικιωμένοι έχουν δικαίωμα στον αθλητισμό. Θα πρέπει να προωθούμε τον αθλητισμό καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, από την παιδική ηλικία μέχρι την ε, ηλικία και νομίζω ότι τρεις ώρες ε, μάθημα γυμναστικής ε, στα σχολεία είναι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλό θα ήταν να έχουμε και ξεχωριστό δημοσιονομικό κεφάλαιο, δημοσιονομική γραμμή για τον αθλητισμό στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για να τηρήσουμε και τη συνθήκη τη Λισαβόνα και την ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για τον αθλητισμό. Ευχαριστώ. Δυστυχώ ε, δεν μπορούμε να παρατείνουμε τη διαδικασία του Catch the Eye, γιατί δεν προλαβαίνουμε, έχουμε και τις παρεμβάσεις ενός λεπτού και πρέπει μέχρι τις 11 να τελειώσουμε. Η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φίσας για την εξαιρετική του έκθεση. Μια έκθεση η οποία είναι ιδιαίτερα συμβατή με τον τρόπο που σκέπτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Αθλητισμό στην Ευρώπη. Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει ήδη κάποιες από τις βασικές ιδέες της έκθεσης. Δεν θα ασχοληθώ με το θέμα των, ε, της σημαίας στις φανέλες και τα λοιπά. Τα μέλη που έθεσαν το θέμα βιάστηκαν να φύγουν κιόλας. Αλλά πάντως ε, υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε στον αθλητισμό και όχι αυτό. το θέμα της βίας σαν παράδειγμα γιατί ξέρετε ότι σήμερα χάθηκαν 70 άνθρωποι λόγω της βίας στα γήπεδα και τραυματίστηκαν άνω των χιλίων. Η βία λοιπόν, το στήσιμο των παιχνιδιών, ο ρόλος των μάνατζερ, όλα αυτά είναι θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε κατεπηγόντως. Προσβλέποντας το μέλλον, ας ε, ενθαρρυνθούμε λοιπόν και από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο πρόγραμμα στον αθλητισμό, το οποίο θα διαθέτει τα μέσα και τα χρήματα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού. Προσβλέπω λοιπόν στη συνεργασία μαζί σας που πιστεύετε όλοι στον αθλητισμό έτσι ώστε να πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε στον αθλητισμό πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Φίσας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Δεν θα ξοδέψω ούτε ένα δευτερόλεπτο για να διαψεύσω μερικές ανακριβείς και ψευδείς παρατηρήσεις. Όποιος δεν ξέρει να διαβάζει τι να πω. Τους παραπέμπω στην έκθεση. Ο αθλητισμός ε, έχει σημαντικό ρόλο στην ε, κοινωνική ένταξη των πιο περιθωριοποιημένων ομάδων. Έχει ε, επωφελή αποτελέσματα στην υγεία, στην απασχόληση, στην οικονομία. Άμεσα ή έμεσα ο αθλητισμός απασχολεί 15 εκατομμύρια ανθρώπους, 5,4% του ενεργού πληθυσμού, με 400, ε, δισεκατομμύρια ε, ευρώ τζίρο του κόσμου, 3,75 δηλαδή του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Είναι τεράστια σημασία του αθλητισμού και χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την υποστήριξή της προς την έκθεση. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Επίτροπο ε, στα διαρθρωτικά ταμεία να, ε, να αφιερωθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία κάποια κονδύλια για τον αθλητισμό. Επίσης, να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες για την υποστήριξη της έκθεσής μου και ευελπιστώ ότι στην αυριανή ψηφοφορία θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Θα ήθελα και εγώ να σας ε, επενέσω για, το, για την εκθέση και να πω ότι όταν ήμουν μέλος ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, συζητούσαμε για τη βία σε αθλητικές εκδηλώσεις ε, στα ποδοσφαιρικά γήπεδα και μερικές εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για το θέμα αυτό θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο μελέτης και να τροφοδοτήσουν τη δική μας συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για την έκθεση το κύριο φύσας και περνάμε στο τελευταίο.